τα κράτη-μέλη οφείλουν εφαρμόσει νομοθεσία στη χώρα τους. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε έτσι η συζήτηση. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι τώρα η κοινή συζήτηση για τη δασική νομοθεσία Καμερούν και Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουμε σύσταση του κυρίου Ζαντού σχετικά με σύναψη θελοντικής συμφωνίας θερικής σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας του Καμερούν και επίσης του ιδίου συντάκτη για σύναψη συμφωνίας θερικής σχέση με τη Δημοκρατία του Καγκό. Του Και υπάρχει και προφορική ερώτηση για τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης που έχει υποβληθεί από περισσότερες ομάδες την οποία επίσης θα συζητήσουμε στο ίδιο σημείο στην κοινή συζήτηση. Δίνω το λόγο λοιπόν πρώτα στον κύριο Ζαντό ως ε, εισηγητή για 6 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να εκφράσω προς όλους τους συναδέλφους τις ευχαριστίες μου για τη δουλειά που έχουμε κάνει μαζί στην υπόθεση αυτή. Οι πολιτικές ομάδες ε, έχουν καταλήξει εκ μέρους του Κοινοβουλίου σε μια κοινή θέση με την υποβολή του ερωτήσεως και του ψηφίσματος που ακολουθεί για τις συμφωνίες εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα για όλους μας. Ξέρετε ότι υποχωρούν τα δάση. Κάθε δύο δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτα χάνουμε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Κάθε χρόνο χάρουμε όλη την έκταση που αντιστοιχεί στην επικράτεια της Ελλάδας σε δασική έκταση. Αυτό έχει τραγικές συνέπειες και για τη βιοπικιλότητα. Χιλιάδες είδη ζώων και φυτών κινδυνεύουν τα δε τροπικά δάση που είναι το περισσότερο σημειώνω ότι εκφράζουν το ίμιση της, Ευρω... της ε, του πλανήτη. Επίσης και ως προς την κλιματική αλλαγή έχει τεράστια σημασία η αποψήλωση των δασών γιατί συμβάλλει σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και επίσης κινδυνεύει η ίδια η επιβίωση 15 πολλών ε, εκατομμυρίων ε, πολιτών ε, του κόσμου που ζουν στα δάση ή από τα δάση. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με υπερεκμετάλλευση. Εδώ έχουμε την πιο σημαντική πηγή της αποψήλωσης και ιδιαίτερα στην περιοχή που μας ενδιαφέρει τώρα, δηλαδή στη λεκάνη του Κόγκο, του ποταμού Κόγκο. μεγάλο ποσοστό των, της ξυλίας που προσφέρεται προς εμπορία ανά τον κόσμο είναι προϊόν παράνομης ε, ξυλοκοπίας. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν συμφωνίες ε, με βάση τη συνένεση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Οργάνωσης ε, Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου όπου Μπορούμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση να εκφράσουμε τι θέσει μα, αλλά μπορούμε μόνο να τι εκφράσουμε με ένα ναι ή με ένα όχι. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε το θέμα, γιατί μπορούμε να επισέλθουμε σε περισσότερε λεπτομέρειε και σε ζητήματα που μα απασχολούν. Και περιμένουμε απαντήσει από εσά, κυρία Επιτροπή, από εκπροσωπείτε την Επιτροπή. Και επίση, έχουμε συμφωνίε οι οποίε επιτρέπουν την ανιχνευσιμότητα τη ξυλία, διαδικασίε ανεξάρτητε, ε, εποπτείας, και παρακολούθηση της ε, πολιτικής των δασών στις ε, χώρες με τις οποίες είναι αυτές συμφωνίες, όπως το Κονκό Μπραζαβίλ και το Καμερούν, εν προκειμένου σήμερα. Ωστόσο, για να επανέλθω σε αυτές τις συμφωνίες και την ερώτηση του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ της ε, νόμιμης και της αϊφόρου ξύλευσης. Ναι, μιλάμε βέβαια για την νόμιμη ξύλευση, αλλά όταν είναι νόμιμη η ξυλία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αντιστοιχεί και σε βιωσιμότητα εκμετάλλευση δασών. Επομένω, η ερώτησή μου προ την Επιτροπή, η πρώτη ερώτηση και κυρία, είναι πώ σκοπεύει η Επιτροπή να εξασφαλίσει την γενική αηφορία για τα δάση, και μην ξεχνάμε το 2011 έχει κηρυχθεί Διεθνέ Έτο Προστασία των Δασών, και λαμβανωμένων υπόψη τα όσα υπόθηκαν στην Εγκόγια, στο Κανκούν πιο πρόσφατα για τον μηχανισμό Red Plus και δεδομένων και των εμπορικών συμφωνιών που συνάπτονται και οι οποίες απελευθερώνοντας μερικές φορές το εμπόριο ξυλίας συμβάλλουν έμεσα στην αποψήλωση των δασών. Και ακόμη θα ήθελα να συμπληρώσω ότι ε, αναμένουμε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, ταξινόμηση, μάλλον την, αναδα... Ε, αναδάσωση και την ε, κατανομή της γης και για τα καύσιμα, για τις εταιρικέ σχέσεις λοιπόν, τις εθελοντικές αυτές σχέσεις συμφωνούμε ιδιαίτερως και υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στο Καμερούν και στην Δημοκρατία του Κόγκο. Ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Αυτές οι, εταιρικές, αυτές οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης λοιπόν έχουν στεφτεί με επιτυχία χάρη στη δική του συμμετοχή. Ε, υπάρχουν επίσης ε, ερωτήσεις όπως έλεγα, αλλά υπάρχουν και αιτήματα. Είστε διατεθειμένος κύριε Επίτροπε να έρχεστε κάθε εξάμηνο από την ε, υπογραφή μιας τέτοιας εθελοντικής συμφωνίας FLECT. Ε, Είσαι διατεθειμένος να έρχεστε κάθε εξάμεινο για να μα για να μας δίνετε έναν λόγο λογαριασμό, έναν απολογισμό του τι έχει γίνει. Γιατί άλλο το τι υπογράφεται και άλλο τελικά το τι γίνεται. Και γι' αυτό θα θέλαμε να έρχεστε και να μας βεβαιώνετε ότι η κοινωνία των ε, πολιτών εξακολουθεί να συμβάλλει σε αυτή, στη λειτουργία αυτών των συμφωνιών ή ειδικά όταν πρόκειται για κράτη τα οποία δεν είναι εύκολο για τον πολίτη να διαμαρτυρηθεί λόγω διαφθορά, Φερρυπίν. Υπάρχουν κάποιε διαδικασίε ή μηχανισμοί για κάποιον φορέα τη κοινωνία των πολιτών, ο οποίο θα μπορούσε να προσφύγει σε εσά και να διαμαρτυρηθεί και να πει ότι τον έχουν βγάλει εκτό παιδιά και δεν, δεν, ακούγεται, δεν ακούγονται οι απόψει του. Και επίση θα θέλαμε τακτική ενημέρωση και για την ε, για τον απόϊχο αυτών των συμφωνιών, για την αποτελεσματικότητά τους και ως προς τα δάση και ως προς το ζήτημα, ως προς το πώς κρίνεται το ζήτημα της νόμιμης ξύλευσης. Και επίσης, για να τελειώσω, θα ήθελα να σημειώσω ότι μας λέτε μένω ότι δεν υπάρχει και προϋπολογισμός, δεν βλέπετε προϋπολογισμός για αυτές τις εθελοντικές με εσωτερικές σχέσεις. Ναι, αλλά οι πολιτικές που θα τις ακολουθήσουν θα χρειαστούν χρηματοδότηση. Πώς, πού θα τη βρείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Και τώρα περνάμε στου συντάκτε ε, τη προφορική ερώτηση. Η κυρία Μπίρτερ για τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Το τροπικό δάσο είναι πολύτιμο στο Καμερούν και στο Κονγκό και πρέπει να καλωσορίσουμε αυτή τη συμφωνία για να αντιμετωπιστεί η βιωσιμότητα της υλοτόμησης εκεί. Οι χώρες αυτές ε, είναι τμήμα, μάλλον το δάσος είναι τμήμα αυτών των χωρών, αλλά είναι και τμήμα του οικοσυστήματος. Συμπεριέχει εκατομμύρια τόνων ε, ε, άνθρακα. Ε, οι κυβερνήσει ολόκληρο τη γη προσπαθεί να χειριστούν ε, τα δάση εδώ και χρόνια και αυτές οι δύο χώρες θα πρέπει να τις συγχαρούμε για το θάρρος τους αλλά και την οραματικότητά τους στην συνυπογραφή αυτών των συμφωνιών. Ένας Θεός ξέρει πώς θα δημιουργήσουμε εμείς ένα σύστημα για τη βιώσιμη διακυβέρνηση της δικής μας υπήρου γιατί εκείνους θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Η προσεκτική διαχείριση μπορεί να μειώσει την ε, εισαγωγή παράνομης ξυλίας. Αυτή τη στιγμή ο όγκος της ξυλίας που παράνομα υλοτομείται και εισάγεται στην Ευρώπη αποτελεί το 1 πέμπτο των προϊόντων ξυλίας στην αγορά μας, παρά τις προσπάθειες χειρισμού και αντιμετώπισης του προβλήματος. Βέβαια, η, η κοινωνία των πολιτών και οι φτωχότεροι άνθρωποι είναι αυτοί που πλήττονται κάθε φορά που λαμβάνονται πιο αυστηρά μέτρα. Γι' αυτό και θα πρέπει να εισακουστούν οι μας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί εκείνοι θα χάσουν τα περισσότερα αν χάσουν τα δάση τους. Η ευρύτατη η εισαγωγή τροπικών, ε, τροπικής ξυλίας οφείλεται στην ε, μεγάλη όρεξη να διακοσμήσουμε τα σπίτια μας. Θα πρέπει ωστόσο να σκεφτούμε ότι τα δάση αυτά όχι μόνο είναι το σπίτι μεγάλο, πολλών ειδών ε, φυτών και ζώων, αλλά και ότι παίρνει πάρα πολλά χρόνια για να οριμάσουν τέτοιου είδους φυτά. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δώσουμε να σταματάψουμε να είμαστε η μεγαλύτερη αγορά για παράνομη ξυλία στον κόσμο. Κάτι τέτοιο μπορεί να σημαίνει ότι η τροπική ξυλία που είναι πολύ ακριβή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας βρει αντίθετο, Όχι μόνο είναι περιορισμένο ο πόρος, αλλά είναι και το μόνο πράγμα που μπορούν να πουλήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Γνωρίζουν την πραγματική αξία του πόρου αυτού. Και χρειάζεται να έχουμε τη δική τους βοήθεια ε, για να επιβληθεί η συμφωνία. Θα πρέπει να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε ώστε να ακούγεται η φωνή τους όταν έχουν ανησυχίες ε, και προβλήματα. Αυτές οι συμφωνίες είναι αμφίδρομες ε, εμείς ε, θέλουμε να είναι καλές και ωφέλιμες για τις χώρες αυτές, καλές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα παρακολουθήσετε την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών και έπειτα θα πρέπει να δούμε και άλλες χώρες, στην Αφρική, την Ασία και την Νότια Αμερική, ώστε να μπορέσουν να υπογράψουν παρόμοιες τέτοιες συμφωνίες όσο γίνεται πιο γρήγορα. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας και με την Επιτροπή για να επιτύχουμε τους στόχους των συμφωνιών αυτών. Ευχαριστώ κύριο Δέβιτ Μάρτιν για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρχίζω με ευχαριστίες προς τον εισηγητή που συνέχισε πάρα πολλά με τους κοιόδες εισηγητές όλους εμάς και τα, οι συμφωνίε αυτές με Γκάνα, Κονγκό, Καμερούν σημαίνει ότι αυτά τα ευάλωτα δάση τώρα καλύπτονται από αυτές τις εταιρικές συμφωνίες και όπως είπαν προλαλήσαντες θα πρέπει να χαιρετήσουμε την υπογραφή των συμφωνιών γιατί είναι μηχανισμός να αντιμετωπιστούν ε, οι τεράστιες ποσότητες της ε, παράνομης Προστατεύουμε τις πρώτες και έτσι ελπίζουμε θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια και θα καταπολεμήσουμε την διαφθορά όσον αφορά την δασική πολιτική που τώρα είναι κάτι το οποίο ενδυμεί ως κακό. Τώρα οι προβληματισμοί μας είναι οι εξής. Πρώτον, ο κίνδυνος δεν έγινε στην πρόθεση αλλά μήπως θεωρούν ότι το ότι θέλουμε να κάνουμε τέτοια ρύθμιση πλαίσιο τόσο ευρέα κλίμακα, ότι θέλουμε να προβούμε σε πάρα πολύ μεγάλη εκτεταμένη υλοτόμηση, το οποίο θα είναι κακό το περιβάλλον. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Θέλουμε συμφωνία που να βοηθά στην διάσωση, στην προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας και συμφωνώ με, τον, ε, με την Επίτροπο ότι χρειάζεται να παρακολουθούμε, θα πρέπει να αναφέρουμε το τι γίνεται. Επίσης, οι θαγενείς λαοί, οι οποίοι τόσο συχνά είναι τα θύματα της μετάλλησης περιβάλλοντος, θα πρέπει και αυτοί να ωφεληθούν. Και η πρόταση προς το, τον λαό κάθε κυβέρνηση είναι να τον προστατεύσει. Θα πρέπει αυτή η υπόθεση και συναντηρηθεί. Θα πρέπει ομένω να φροντίσει και η Κομισιόν να τηρηθούν τα επισχημένα. Και σε όλε τι χώρε και κύριε στο Κονγκό αυτή η νομοθεσία να αποτελέσει πραγματικότητα. Ε, επίσης θα πρέπει οι πόροι να δοθούν εκεί που έχει πραγματικά υιοθετηθεί το νομοθέτημα, γιατί χωρίς τους πόρους δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εφαρμογή νομοθεσίας. Επαναλαμβάνουμε, χρηματοδοτικά πακέτα δεν συνδέονται άμεσα με τη συμφωνία. Εμείς, το Συμβούλιο, θα κάνουμε την ε, αναγκαστική δέσμευση πόρων στον προπολογισμό τους, ώστε να βοηθεί η εφαρμογή των ε, νομοθετημάτων αυτών. Και έτσι να έχουμε νόμιμη ξυλία που να εισάγουμε. Μπορούμε να παρέχουμε τεχνικές συμβουλές σε αυτούς που επιτόπου ασχολούνται με τον κλάδο και να υπάρχουν απαραίτητοι πόροι, ούτως ώστε να γίνει παντού αυτή όλη η υποπτία. Και άρα μετά από το νομοθετικό πλαίσιο έχουμε και το χρηματοδοτικό πλαίσιο. Παραλαμβάνω, πρόκειται για αξιολόγηση συμφωνίε. Όπω όλε όμω, όλα θα εξαρτηθούν από την καλή πίστη, την επαγρύπνηση, τι θα κάνουν ε, οι κυβερνήσεις, οι λαοί, <clears throat> αυτοί να εξασφαλίσουν το ότι και στην πράξη θα αποδώσει αυτή η νομοθεσία. Να γίνει καλύτερη διαχείριση επομένως, τόσο ώστε να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε το ρεύμα. Άρα η Κομισιόν θα πρέπει να επαγρυπνεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τζο δύο λεπτά. Συμφωνώ πάρα πολύ με τον Γιάννη στη γενική του προσέγγιση. Εγώ καλωσορίζω οποιαδήποτε συμφωνία που θα εγγυηθεί την προστασία των ε, δασών στον πλανήτη. Αυτό σημαίνει προστασία των ε, αυτοχθόνων κατοίκων των δασών, που είναι καθώς και την πλειοψηφία των πολιτών των εν λόγω χωρών. Η, το Κονγκό και το Καμερούν έχουν πολύ καταπιεστικές ε, κυβερνήσεις εντωμεταξύ. Το Καμερούν είναι πολύ ψηλά δε στον δίκτυο της διαφθοράς και το Κονγκό ε, είναι γνωστό για την ε, πολύ κακή μεταχείριση κάποιων λαών που κατοικούν εκεί, ιδιαίτερα των πυγμαίων που κατοικούν στη χώρα. Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών είναι μέσα στη διαφθορά και η υποψήλωση είναι τεράστιο σπόρος για τις ζωές ε, των αυτοχθόνων των περιοχών αυτών και γι' αυτό και η Γκουε ζητά από τη ζητά οι εταιρείε υλοτόμηση να είναι δημόσιες εταιρείε και να ε, στο ψήφισμά μας τονίζουμε επίσης ότι η παράνομη υλοτόμηση σχετίζεται με τα επίπεδα φτώχειας των λόγω χωρών. Μπορεί να τους βοηθούν δηλαδή στον κόσμο να μπορέσουν να ζήσουν γιατί διαφορετικά θα υπέφεραν από πείνα Και βέβαια αυτό το θέμα δεν πρόκειται να ρυθμιστεί από τις τοπικές ε, διεφθαρμένες ελίτ, ούτε από τις μεγάλες ε, διεθνείς, ε, μάλλον πολυεθνικές εταιρείες. Μόνο αν ο κόσμος μπορέσει να αναλάβει, ο λαός μάλλον των χωρών αυτών μπορέσει να αναλάβει τη διαχείριση των δασών τους και αν εμπνευστούν από τους αδερφούς τους και τις αδερφές του την Ισία στο δικό τους αγώνα κατά μιας διεφθαρμένης δικτατορίας τις τελευταίες εβδομάδες θα υπάρξει κάποια λύση. Ο κύριος Κάσπερ για δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, έχουν ξεκινήσει τα κράτη τα οποία εξάγουν σκληρή τροπική ξυλία να συνάπτουν θεωρητικέ συμφωνίε εταιρική σχέση με τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη διεκδικεί και ε, σωστή διαχείριση των δασών και ε, ένα σύστημα ανιχνευσιμότητας ταυτόχρονα και της νομιμότητας της ξυλίας που έχει υλοτομηθεί. Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως είναι η βελτίωση της διαφάνειας και η αποτροπή των, ε, της αποψήλωσης των δασών. Σε αυτό μπορούν να συμβάλλουν αυτέ οι θεωρητικέ συμφωνίε εταιρική σχέση εφόσον βελτιωθούν και τροποποιηθούν σχετικά. Επίση, η ανάπτυξη των ε, ικανοτήτων στι χώρε παραγωγή αυτή τη ξυλία, ιδιαίτερα με ένα σύστημα και προέλευση και ε, νομιμότητα, ελέγχου δηλαδή προέλευση και νομιμότητα, είναι πολύ σημαντική. Αυτέ οι εθελοντικέ εταιρικέ ε, σχέσει θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουν σαν, κύριο, σαν κύρια πηγή έπνευση στην βούληση να τεθεί ένα πέρα στην εμπορία προϊόντων ξυλία που προέρχονται από παράνομη, παράνομη ηλιοτομία και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, δεν μπορούμε να δεχθούμε την καταστροφή των τροπικών δασών, τα οποία έχουν τόσο μεγάλη σημασία για τον πλανήτη μας. Είναι λοιπόν ένα μικρό βήμα, αλλά ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτές οι θελοντικές συμφωνεστερικές σχέσεις ε, προς την ορθή κατεύθυνση. Ευχαριστώ ε, όλους τους συντάκτες που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Συμφωνώ με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα και ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτές τις συμφωνίες. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο Επίτροπος Πίμπαλξ, παρακαλώ. Πρόεδρε. Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή κύριο Ζαντό για την υποστήριξή του στι ε, θελοντικέ αυτέ εταιρικέ συμφωνίε για την ε, διαχείριση των δασών στο Κονγκό και στο Καμερούν. Ελπίζω πως θα ακολουθήσετε τις συστάσεις τους για συγκατάθεση προς αυτή τη συμφωνία, στο να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι, αλλά όσο και οι ε, χώρε εταίρε να εγκρίνουν αυτή τι συμφωνίε, γιατί η παράνομη υλοτομία είναι πρόβλημα για όλους. Η νόμιμη υλοτομία είναι μόνο το, η κορυφή του παγόβουνου. Μιλάμε βασικά την αρχή μιας συνεργασίας για τη βιώσιμη διαχείριση των βασικών πόρων. Και για να απαντήσω σε μια από τις συστάσεις του εισηγητή, ναι, να πω ότι είμαι έτοιμος να έρχομαι κάθε έξι μήνες ή όποτε με καλείτε και να παρακολουθώ την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Είναι αλήθεια πως πρόκειται για δέσμευση. Υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά είναι ο μόνος τρόπος κατά τη γνώμη μου να κατευθυνθούμε προς την βιώσιμη διαχείριση αυτών των πόρων. Αν δεν το κάνουμε αυτό, μόνο με δηλώσεις δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα. Για τις χώρες εταίρους υπάρχει μεγάλη δέσμευση και διάθεση. Πολύ σημαντικό είναι ότι, ε, είναι πολύ, ε, ε, από, ότι ζημιώνονται από την παράνομη υλοτομία. Κάθε χρόνο 10 με 15 δις δολάρια χάνονται λόγω της παράνομης υλοτομίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα ζημιογόνο για τους αυτόχθονες ε, της περιοχής αλλά και για την κλιματική αλλαγή. Είναι πολύ σημαντικό εξάλλου να τονίσουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές για τα τροπικά, τροπική ξυλία σημαίνει ότι και η δική μας προσέγγιση είναι πολύ σημαντική για το πώς αντιμετωπίζεται το θέμα. 20% του το τροπικής ξυλίας φτάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προέρχεται από, παράνομη, από παράνομες πηγές. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι η μόνη μας ε, πόρη, ε, ότι θα χρησιμοποιούμε μόνο νόμιμο, νόμιμη ξυλία. Ταυτόχρονα οι κλιματικές αλλαγές είναι ανησυχία όλων και η προστασία των δασών κάπου θα πρέπει να ξεκινήσει. Είναι απλό να λέμε ότι πρέπει να πληρώσουμε για να προστατευτούν τα δάση. Είναι απλό, αλλά για να το εφαρμόσουμε χρειάζεται μεγάλη δέσμευση και από τις δύο πλευρές. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ένα-δυο ερωτήσεις που μου ετέθησαν για την επιβολή και την εφαρμογή οι συμφωνίε προβλέπουν κοινή επιτροπή για την εφαρμογή που παρακολουθεί την εφαρμογή τη συμφωνία. Επίση, θεσπίζεται ανεξάρτητο έλεγχο που θα αναλύει την αποτελεσματικότητα και την ε, απόδοση του συστήματος. Ετήσιες εκθέσεις θα δημοσιεύονται και θα είναι διαθέσιμες φυσικά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, μέσω της προετοιμασίας για αυτή την εθελοντική συμφωνία έχουμε ήδη ε, εμπλέξει τις, ε, τους τοπικούς πληθυσμούς. Μέχρι τώρα είχαν αφαιθεί τελείως εκτός της διαδικασίας. Γι' αυτό και συμφωνήσαμε μέσω αυτών των συμφωνιών ότι θα δημιουργηθούν ε, επιτροπές με μεγάλη συμμετοχή και των ε, τοπικών ε, πληθυσμών. Επίσης, ο ανεξάρτητος ελεγκτής θα έχει πρόσβαση και θα βασίζεται σε πληροφορίες από μεγάλη ποικιλία πόρων και από την κοινωνία των πολιτών, αλλά και από τις τοπικές κοινότητες. Ανάμεσα στο 2002 και το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε με 544 δις ευρώ για τη δασοκομεία στον αναπτυσσόμενο χώρο. Ορισμένα από αυτά τα χρήματα πήγαν σε συγκεκριμένε χώρε. Η Κομισιόν έχει δαπανίσει 35 εκατομμύρια για να υποστηρίξει το ΦΛΕΚΤ γενικότερα και 35 εκατομμύρια επιπλέον ανάμεσα στο 2011 και το 2013 προβλέπονται. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι τα κράτη-μέλη κάνουν δικές τους ε, συμβολές. Έχουμε επίσης αφιερώσει ανθρώπινους πόρους για την εφαρμογή των ΦΛΕΚΤ. Εγώ έχω 7 υπαλλήλους που ασχολούνται με αυτό το θέμα και συνεργάζονται στενά με το Ευρωπαϊκό Δασοκομικό Ινστιτούτο και με τις Εθνικές Δασοκομικές εταιρείε. Επίσης έχουμε κάποια επιπλέον βοήθεια από το πρόσφατο κανονισμό που υιοθετήθηκε για την παράνομη υλοτόμηση ένα πρόγραμμα κλειδί ε, δράσης ε, το οποίο θα συμπληρώσει τις ε, θελοντικές συμφωνίες εταιρική σχέσης. Η πρόσφατη συμφωνία στο Κανκούν για τη μείωση των εκπομπών λόγω αποψήλυσης ή υποβάθμισης των δασών θα διευκολύνει περαιτέρω στήριξη από την Κομισιόν Προ τι αναπτυσσόμενες χώρες. Η μελλοντική μας ε, δουλειά για την διακυβέρνηση των δασών μέσω θελοντικών συμφωνιών εταιρική σχέση, ε, θα προβλέπει συνεργασία με την κυβέρνηση σε σεβασμό των τοπικών ε, κοινοτήτων και των αυτοχθόνων ηθαγενών. Συμφωνώ με το σχέδιο ψηφίσματος ότι η Κομισιόν θα πρέπει να παρακολουθεί ε, και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας διαβεβαιώ. Είναι στο επίκεντρο προσοχή μας όσον αφορά αυτές τις χώρες. σα εξασφαλίζω ότι θα καταπολεμήσουμε την διαφθορά που είναι ένα από τα θέματα τα οποία μας καίνε και πρόκειται να το συζητήσουμε τι χώρε αυτέ, Αλλά όμω θέλω να τονίσω για να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο απετέλεσε αιτία ενθάρρυνση. ότι δηλαδή θεωρούν δεσμευμένες αυτές οι χώρες ε, οι εταίροι μας. Και ακριβώ ξέρουν ότι υπάρχουν κάποιε αδυναμίες και ότι έτσι θα προστατεύσουν τελικά ε, το, το, το, Όμως αυτό είναι μόνο η αρχή. όμω ακριβώς πρόκειται για μια αφετηρία που είναι κοινή και όλα αυτά ε, φυσικά θα τα αναφέρουμε το πώ προχωράει η εφαρμογή. Όμω πρέπει να σα ξαναπώ ότι δεν έχουμε κάνει κανένα λάθο βήμα. Έχουμε κάνει βήματα μόνο προ σωστή κατεύθυνση και ε, όντω υπάρχουν κίνδυνοι, τους δεν ε, έχουμε έτοιμε λύσει, αλλά πρόκειται για ένα βήμα, το οποίο μα έχει κάνει περήφανος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε, Πρόεδρος. Πρώτα-πρώτα να με συγχωνρώνουν οι δύο συνάδελφοι που τους διέκοψα εν τη ροή της ομιλίας τους αλλά μόλις ε, αντικατέστησε τον προηγούμενο αντιπρόεδρο